Ε, ε, Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ζητήσω από τις τεχνικές υπηρεσίες να κάνουμε μία δοκιμή για να δούμε κατά πόσο λειτουργεί το ηλεκτρονικό σύστημα ως προς τις ηλεκτρονικές μας ε, κάρτες, διότι μου είπαν από τα γραφεία μας ότι με αυτό το νέο σύστημα δεν λειτουργούν όλες οι κάρτες. Θα ήθελα λοιπόν να κάνουμε μία δοκιμή, να βάλετε την κάρτα σας για να δούμε κατά πόσο εμφανίζεται το όνομά σας. Εάν ισχύει κάτι τέτοιο, αυτό σημαίνει ότι λειτουργεί το σύστημα. Εάν δεν εμφανιστεί το όνομά σας, στον χώρο που προβλέπετε, τότε αλλάξτε θέση και προσπαθήστε να δείτε κατά πόσο δίπλα λειτουργεί το σύστημα. Θέλετε το λόγο. Ο κύριος Άτκινς. Εντάχει θα κάνω ό,τι μου πείτε, αλλά για το μέλλον να ξέρετε ότι δεν λειτουργεί στη δική μου θέση και επειδή θα κάθομαι αρκετά συχνά ελπίζω να λειτουργεί στο μέλλον. Σας ευχαριστώ όλοι. Συμφωνούμε με τον κύριο Άτκινς, διότι το σύστημα πρέπει να καταστεί λειτουργικό. Αλλά θα ήθελα να σας ζητήσω για αυτή τη φορά να προσαρμοστούμε κάπως. Εάν δεν λειτουργεί η κάρτα σας στη δική σας θέση, και αν αφού την εισαγάγετε δεν ε, αναγράφετε το όνομά σας, θα πρέπει να το δοκιμάσετε δίπλα, κάπου δίπλα, μέχρι ότου δείτε το όνομά σας, για να είμαστε σίγουροι ότι λειτουργεί. Εάν έχετε εισαγάγει την κάρτα, τώρα θα κάνουμε τη δοκιμή. Λοιπόν, ψηφίστε για να δούμε αν λειτουργεί το σύστημα και για να επαληθεύσουμε τον αριθμό των ε, παρόντων. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Είμαστε 33 ε, παρόντες. Ποιοι έχουν προβλήματα. Εάν έχετε πρόβλημα, δοκιμάστε δίπλα. Κάντε μια άλλη δοκιμή. Κύριε Τάνοκ, μας το κοινοποίησατε. Κάντε αυτή τη δοκιμή δίπλα. Εντάξει, λειτουργεί. Κύριε Τάνοκ, πηγαίνετε δίπλα, το ξαναείπα. Ε, σε Εάν εμφανίζεται το όνομα, πάει να πει ότι λειτουργεί. Και μετά θα πρέπει να εισαγάγεται την κάρτα σας. Σας κάνουμε άλλη μια δοκιμή. Έχετε εισαγάγει την κάρτα στο μηχάνημα. Πράσινο, κόκκινο ή λευκό. Δοκιμάστε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Κάνατε τη δοκιμή όλοι. Εντάξει. 49 Ψήφισαν 49, 36 και 6 και 7 αποχέ. Υπάρχει κάποιος που θα ήθελε να κοινοποιήσει ότι δεν λειτουργεί το σύστημα στη θέση του. Εντάξει, φαίνεται πως όχι, εντάξει. Μπορούμε να αρχίσουμε λοιπόν με τις ψηφοφορίες. Εάν συμφωνείτε, αρχίζουμε με την ψηφοφορία του προϋπολογισμού τμήμα τρίτο. Η συγγήτρια Νέιτς. Ας αρχίσουμε με μία unblock ψηφοφορία από την τροπολογία 5021 μέχρι την 5016. Υπέρ. διανατάσεως κατά αποχές εγκρίνεται. Unblock. 5036 της εισηγήτριας υπέρ διανατάσεως κατά αποχές εγκρίνεται. 50-37 υπέρ. Σηκώστε το χέρι παρακαλώ. Κατά. Εγκρίνεται. 50-38 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 50-28 υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Μάλλον όχι, φαίνεται ότι απορρίπτεται. Καλύτερα να ελέγξουμε. Λοιπόν, αρχίζει η ψηφοφορία επί της τροπολογίας 50-28 της εισηγήτριας. Αρχίζει η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Σας παρακαλώ να ψηφίσετε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. Ψήφισαν 54, 25 υπέρ, 27 κατά, συν ένας κατά, άρα 28, δύο αποχές, άρα απορρίπτεται η τροπολογία. Είσαστε υπέρ ή κατά. Λειτουργεί. Εντάξει. Όπως και να έχει απορρίπτεται. Γιατί είμαστε κάτω από το κατόφλι και ο κύριος Κάτσιν υπέρ. 27 υπέρ 28 κατά. Α, 28 υπέρ 29 κατά. Άρα μεταξύ ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και διαχειρός είμαστε 28 έναντι 29, άρα απορρίπτεται. 5.008 υπέρ. Κατά. 50.67 υπέρ. Κατά. 50.11 υπέρ. Κατά απορριπτεται 5012 υπέρ κατά 5027 50-27 της εισηγήτριας υπέρ κατά εγκρίνεται. 5.009 όπου έχουμε ξεχωριστή ψηφοφορία. Ψηφίσουμε μόνο το δεύτερο τμήμα. Ποιοι τάσσονται υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα. 50-51. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 50-49. Υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Κύριε Σαλαφράνκα, ζητήσατε το λόγο, έχετε το λόγο. Δεν ξέρω κατά πόσο υπήρξε κάποια παρεξήγηση λόγω ρυθμού ως προς το 50-51. Είπα χθες ότι αποσύρω το πρώτο τμήμα και άρα ε, αναφερόμαστε μόνο στα σχόλια και σε τίποτα παραπάνω. Αυτό είπα χτες. Νομίζω ότι ψηφίσαμε όπως ορίζει και ο κατάλογος ε, ψηφοριών. Only remarks, δηλαδή μόνο τα σχόλια. Άρα έχετε απόλυτο δίκιο. 50-49 δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Μάλλον εγώ δεν είδα καλά. Ας προβούμε σε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αρχίζει η ψηφοφορία, επαλήθευση, επαλήθευση, 50-49. Ψηφίσατε όλοι. Σας παρακαλώ, ψηφίστε. Tutti hanno Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Ψήφισαν 56, 23 υπέρ, 32 κατά. Μία αρα απορρίπτεται. 50-52 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός 1. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Άρα εκπίπτει η επόμενη 50-73. 50-69 ψηφίζουμε τώρα. Υπέρ παρακαλώ κατά, απορρίπτεται. 50-29 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 50-26 της εισηγήτριας υπέρ, υπέρ, επαναλαμβάνει ο πρόεδρος. Α, όχι, όχι, καταπίπτει, καταπίπτει και αυτή. Η 5029 δεν εγκρίθηκε, άρα ψηφίζουμε την 5026. Θα εξέπιπτε μόνο αν εγκρινόταν η προηγούμενη. Άρα ψηφίζουμε την 5026. Διανατάσεως υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε unblock από την 5000 μέχρι την 5065. Καλά τα λέω, λέει ο πρόεδρος. Υπέρ. Ναι, βλέπω ότι ψηφίζουμε αν μπλοκ. Υπέρ. Α, όχι, λέει η γραμματεία. Ε, μεμονωμένα πρέπει να τις ψηφίσουμε, ορίζει η γραμματεία. Με συγχωρείτε, λέει ο πρόεδρος. Κύριε Σαλαφράγκα, έχετε το λόγο. Εμείς τα προτιμούσαμε να μην γίνει ψηφοφορία unblock, διότι υπάρχει διαφοροποίηση ως προσωρισμένα τμήματα και θα θέλαμε να ψηφίσουμε πρώτα την 5.000 και μετά τη συνέχεια Allora, Η θέση του κυρίου Σαλαφράνκα και νομίζω ότι είστε εκπρόσωπος του ΕΛΚ είναι να ψηφίσουμε την 5.000 χωριστά και τις υπόλοιπες αμπλόκ ζητάτε ή την καθεμία χωριστά. Α, όλες ξεχωριστά. Την καθεμία χωριστά. Σε αυτή την περίπτωση Εάν μια πολιτική ομάδα θέλει να ψηφιστούν ε, μεμονωμένα, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Πρέπει να λάβω υπόψη την ε, κατάσταση και θα πρέπει να ψηφίσουμε την καθεμία ξεχωριστά. Αυτό προβλέπει ο κανονισμός. Δυστυχώς θα χάσουμε λίγο περισσότερο χρόνο. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο. Λοιπόν, 50-53, λέει ο πρόεδρος. Α, με συγχωρείτε, λέει ο πρόεδρο. 5.000. 5.000. Υπέρ. Βοτι... Κατά. Απορρίπτεται. 50-53. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 5.001 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 50-54 υπέρ κατά 5068 υπέρ κατά εγκρίνεται. 5.002 υπέρ κατά απορρίπτεται. 50-57 υπέρ κατά εγκρίνεται. 50-58 υπέρ κατά εγκρίνεται 50.003 υπέρ κατά απορρίπτεται 50.59 υπέρ κατά εγκρίνεται 5.004 υπέρ κατά απορρίπτεται 50.60 υπέρ κατά εγκρίνεται. 5.005 υπέρ κατά απορρίπτεται. 50.62 υπέρ κατά εγκρίνεται. 50.63 υπέρ κατά εγκρίνεται. 50.64 υπέρ κατά εγκρίνεται. 5.006 υπέρ κατά απορρίπτεται 5.065 υπέρ κατά εγκρίνεται δεν ε, ζητώ τους απέχοντες για να το δούμε πιο γρήγορα Εάν κάποιο κάποιος το επιθυμεί διακάως, μετά την έγκριση, την απόρριψη, μπορεί να το ζητήσει. Θα καταγράψω την αποχή αν υπάρχει. Λοιπόν, 50-13 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 50-41. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 50-42 υπέρ κατά εγκρίνεται. 5.007 μόνο τα σχόλια υπέρ κατά εγκρίνεται. 50-33 της εισηγήτριας υπέρ κατά εγκρίνεται. 50-50 υπέρ κατά εγκρίνεται. 50-55 υπέρ κατά εγκρίνεται 50-34 της εισηγήτριας υπέρ κατά εγκρίνεται 50-70 υπέρ κατά απορρίπτεται 50-30 υπέρ κατά απορρίπτεται. Στην 50 68 έχουμε ξεχωριστή ψηφοφορία. Για το πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, νομίζω ότι εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Α, θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο, εντάξει. Αρχίζει η ψηφοφορία. Η ηλεκτρονικά για το πρώτο τμήμα. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Α, όχι, ας περιμένουμε. Ξαναρχίζουμε. Στο προς το πρώτο τμήμα για την 5068 αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Ψήφισαν 62, 43 υπέρ, 19 κατά. Καμία αποχή. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. κατά εγκρίνεται. Μα με συγχωρείτε, ήταν σαφές. Εντάξει, εντάξει, τι να κάνω. Εντάξει. Αρχίζει η ψηφοφορία για το δεύτερο τμήμα της 5068. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας.

κατά εγκρίνεται. 50-14 υπέρ κατά απορρίπτεται. 50-43 της εισηγήτριας υπέρ κατά εγκρίνεται. 50-72 υπέρ κατά Απορρίπτεται. 50-17 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 50-23. Διότι 50 είναι παρόμοια. Ψηφίσουν 50-23 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 50-22 υπέρ κατά εγκρίνεται. Εάν συμφωνείτε, μπορούμε να ψηφίσουμε από κοινού την 44, 45, 46, διότι είναι η αποκατάσταση των, του αρχικού ποσού εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Άρα ψηφίζουμε μπλοκ την 44, 45 και 46 υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται. 50-35 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 50-24 της εισηγήτριας υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Περνάμε τώρα ε, στο σχέδιο γνωμοδότησης και έχουμε ένα κατάλογο ψηφοφορίας που αρχίζει με την 1 υπέρ, υπέρ παρακαλώ, Είσαστε έτοιμοι. Λέζινγκ, Μάιερ, ψηφίζουμε επί της 1. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Απορρίπτεται. 2. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 3. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ κατά ε, απορρίπτεται νομίζω πέντε, υπέρ κατά εγκρίνεται έξι, υπέρ κατά εγκρίνεται έπτα, υπέρ κατά εγκρίνεται 8 υπέρ κατά εγκρίνεται 9 υπέρ κατά εγκρίνεται 10 υπέρ κατά Νομίζω ότι πρέπει να γίνει ηλεκτρονική επαλήθευση. Ας ψηφίζουμε τις 10 Orden. Αρχίζει ηλεκτρονική ψηφοφορία. Orden. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Ψήφισαν 64, 27 υπέρ, 36 κατά, άρα απορρίπτεται. Τροπολογία 11. Διανατάσεως υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται νομίζω. 12. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 13. Επειδή δεν εγκρίθηκε η 12. Υπέρ της 13. Κατά. Εγκρίνεται. Άρα έχουμε την ηλεκτρονική ψηφοφορία επί της γνωμοδότησης. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Με συγχωρείτε, λέει ο πρόεδρος. Θα πρέπει να ξαναψηφίσουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την πρόταση. Ψηφίσατε όλοι. Δεν λειτουργεί το σύστημα. Ε, υπάρχουν άλλοι που έχουν ε, πρόβλημα με τις κάρτες τους. Πείτε μας λοιπόν. Με συγχωρείτε. Όταν πιέζω το πράσινο αναγράφεται το άσπρο φαίνεται το άσπρο. Θα σας ε, ζητούσα να ψηφίσετε διανατάσεως. Δεν μπορούμε να σας πούμε να μετακινηθείτε. Λειτουργεί αλλά λάθος. Ακόμα χειρότερα λέει ο πρόεδρος. Λοιπόν, υπέρ. Άρα, θα, ωραία, θα ψηφίσουμε, θα προσθέσουμε μάλλον την ψήφο σας. 50 συν 1. 51 6 κατά 5 αποχές. Ωραία, να συγχαρούμε την εισηγήτρια, την κυρία Νέιτς. Ήταν επίπονο το έργο της. Είχαμε και μερικά μικροατυχήματα, αλλά τι να κάνουμε. Ο κύριος Πέτερλε ζήτησε να παρέμβει πριν από την ψηφοφορία της εκθέσεις τους. Κύριοι συνάδελφοι, ε, θα ήθελα να σας πω ότι προσπαθήσαμε να συμπεριφερθούμε οικολογικά και ως προς την 38 που αποσύρθηκε την τροπολογία αυτή δεν ε, προτείναμε ένα νέο κατάλογο ψηφοφοριών. Θα ήθελα να προσθέσω ότι θα γίνει μια διόρθωση τεχνικής φύσης σε σχέση με την αιτιολογική σκέψη 6, διότι υπάρχουν 27 κράτη-μέλη που έχουν κυρώσει αυτή τη συμφωνία. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτές τις διευκρινήσεις. Μπορούμε να προχωρήσουμε τώρα ως προς ε, το σχέδιο ε, ψηφίσματος συνεργασία με το Τατζικιστάν. Αρχίζουμε με την 24, τροπολογία 24, υπέρ παρακαλώ. 24, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 25, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 26 του εισηγητή υπέρ κατά εγκρίνεται 27 Χάουταλα, Μπραντερ και άλλων υπέρ κατά εγκρίνεται τροπολογία 28 υπέρ κατά εγκρίνεται τροπολογία συμβιβασμού 1 υπέρ κατά εγκρίνεται, άρα καταπίπτει η 29 και, και η 30. Ψηφίζουμε την τροπολογία 31 του εισηγητή υπέρ παρακαλώ. Κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 34 υπέρ. Κατά Απορρίπτεται. Τροπολογία 32. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 33. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 36. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 35. Υπέρ κατά εγκρίνεται 37 υπέρ κατά εγκρίνεται 38 αποσύρθηκε περνάμε στην 39 υπέρ κατά εγκρίνεται 40 υπέρ κατά εγκρίνεται Εάν κάποιος θέλει να απόσχει να μου το πει για να καταγράψω την ψήφο του. Δεν του αναφέρω για να κινηθούμε πιο γρήγορα. Περνάμε στην 41 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 42. Υπέρ. Κατά εγκρίνεται 43 υπέρ κατά εγκρίνεται 44 υπέρ κατά εγκρίνεται 46 ε, υπέρ κατά εγκρίνεται 45 υπέρ κατά νομίζω ότι απορρίπτεται 47 υπέρ κατά εγκρίνεται 48 υπέρ κατά εγκρίνεται 49 υπέρ κατά εγκρίνεται Τροπολογία συμβιβασμού υπαριθμών 2. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Καταπίπτει η 50 και 51. Καταπίπτουν. Μετά από την έγκριση της τροπολογίας συμβασμού υπαριθμών 2. Ψηφίζουμε λοιπόν την 52 του εισηγητή υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 53 καταπίπτει. 54 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Εδώ υπάρχει μία προφορική τροπολογία που δεν επαναλαμβάνω. Την βρίσκεται καταγεγραμμένη στον κατάλογο ψηφοφοριών. Είναι η 55 την οποία και ψηφίζουμε υπέρ κατά εγκρίνεται 56 υπέρ κατά εγκρίνεται 57 υπέρ κατά εγκρίνεται 1 υπέρ κατά νομίζω ότι έχει απορριφθεί Θέλετε να ελέγξουμε. Δεν είμαι και απόλυτα ε, σίγουρος. Από ευσυνειδησία και μόνο ας κάνουμε ε, μια ηλεκτρονική επαλήθευση. Για την τροπολογία υπαριθμών 1. Ανοίγει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Εγώ ψηφίζω υπέρ. Να το ξέρετε. Πέρας. 26 συν 1 υπέρ, 27, 33 κατά, άρα απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη Β, 2 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία του ησυχητή εδώ, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Άρα καταπίπτουν οι 3 και 4. Μετά από την έγκριση αυτή ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 5 υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ κατά απορρίπτεται. 6 ε, συγγνώμη υπέρ κατά απορρίπτεται. 8 του εισηγητή υπέρ κατά εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά εγκρίνεται. 11 υπέρ κατά απορρίπτεται. 10 υπέρ κατά Απορρίπτεται. Α, με συγχωρείτε, λέει ο πρόεδρος. Εγκρίνεται. 12. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 13. Υπέρ. Α, συγγνώμη, καταπίπτει, διότι εγκρίθηκε η 12. Τροπολογία 14. Υπέρ. Κατά εγκρίνεται 15 υπέρ κατά εγκρίνεται 16 υπέρ κατά εγκρίνεται 17 υπέρ κατά εγκρίνεται 18 του εισηγητή υπέρ κατά εγκρίνεται. 19 το εισηγητή υπέρ κατά εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά απορρίπτεται. 22 υπέρ κατά Εγκρίνεται 23 υπέρ κατά εγκρίνεται. Με ηλεκτρονική ψηφοφορία έχουμε και την τελική ψηφοφορία ως προς την πρόταση έκθεσης. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψήφισαν 58, 51 υπέρ. Ε, εσείς τι ψηφίζετε. Απλώς να... Α, είσαστε υπέρ, ωραία. 51 συν, συν 1. Α, 52 υπέρ. Α, 53 υπέρ. 7 κατά και καμία αποχή. Ένα σχόλιο εκτός μικροφώνου. Una richiesta di intervento, non ho capito. Θέλετε το λόγο. Qualcuno vuole intervenire. Ποιος θέλει το λόγο. Prego, ha la parola, collega. Prego. da questo vai za. Non, lei ha, Ha votato a favore. Ψηφίσατε υπέρ, εντάξει, ωραία. Tale dei voti a favore è 51 per voto elettronico e 3 51 υπέρ με ηλεκτρονική και 3 χειροκίνητα, α το πούμε έτσι, λέει ο πρόεδρος. 54 συνολικά. Να συγχαρούμε λοιπόν τον εισήγητη. Άρα ψηφίζουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία την πρόταση γνωμοδότησης χωρίς τροπολογία. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την πρόταση γνωμοδότησης. Εάν δεν λειτουργεί το μηχάνημά σας, να μας το κοινοποιήσετε για να ξέρουμε πώς ψηφίσατε και να σας συμπεριλάβουμε. Εσείς ε, τάσεστε υπέρ. Λοιπόν, υπέρ, υπέρ, μιλώ για αυτούς που δεν έχουν την κάρτα ή των οποίων η τον οποίο η καρτα δεν λειτουργεί. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ. Τέσσερις. Πέρας. 51 συν 4, 55, 7 κατά μία αποχή, άρα η πρόταση γνωμοδότησης εγκρίνεται. Να συγχαρούμε τον εισηγητή και τελειώσαμε με τις ψηφοφορίες. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή και όπως σας είχα πει χτες λάβαμε υπόψη τις προτάσεις Λούνατσεκ και άλλων και έτσι ο κύριος Μόραν και η κυρία Αρνό μπορούν να μας ενημερώσουν για την κατάσταση Ο κύριος Μωράν είναι υπεύθυνο για θέματα Ασίας και η κυρία Αρνό θα μας μιλήσει για το Αφγανιστάν. Άρα θα δώσω το λόγο στον δόκτωρα Μωράν καταρχήν. Έχετε το λόγο για την κατάσταση στο Αφγανιστάν. Κύριε Πρόεδρε, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο απόψεις στην παρέμβασή μου. Θα ζητήσω από τον συνάδελφο Αρνό να μιλήσει για την κατάσταση επιτόπου. Λοιπόν, το πρώτο θέμα που θέλω να δούμε είναι οι πιθανές εξελίξεις των επομένων μηνών. Εδώ πρέπει να πούμε καταρχήν ότι όποια και αν είναι η έκβαση, οι εκλογές έπαιξαν το ρόλο τους για να αλλάξουν λίγο την ισορροπία μεταξύ εθνοτήτων στο Αφγανιστάν. Ο δόκτωρ Αμπτάλα έκανε στεναρή εκστρατεία. Ε, μπορεί να θέλουν περισσότερα υπουργεία, ε, μεγαλύτερη ισχύ στο μέλλον. Σημαντικό είναι να τα ξέρουμε όλα αυτά, να εργαστούμε με όλους τους εκπροσώπους, ούτως ώστε ε, να αποφορτήσουμε συναισθηματικά τα πράγματα και να είναι ρεαλιστικές οι λύσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό μετά τη γνωστοποίηση, την κοινοποίηση του εκλογικού αποτελέσματος να ξέρουμε ότι θα είναι μια ε, επαρκής ικανή διοίκηση η οποία θα ε, αφοσιωθεί στην αναβάθμιση της βιωσιμότητας του Αφγανιστάν με μια δίκαιη ε, και συνεπή κοινωνία. Ο ρόλο κλειδί ε, έπαιξε η Επιτροπή Εκλογικών Ενστάσεων, πολύ σημαντικό, με την πλήρη υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας και η Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια ε, παίζει ρόλο, είναι κέρια αυτή η διαδικασία, θα, θα επανέλθουμε αργότερα. Εις ό,τι αφορά το μέλλον, θα θυμάστε ότι τον Ιούνιο το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων εκάλεσε την Κομισιόν, τη Γραμματεία του Συμβουλίου και την Προεδρία να εξετάσουν την κατεύθυνση που ακολουθούμε στο Αφγανιστάν και να υποβάλει συστάσεις το φθινόπορο σχετικά με το τι θα πρέπει να γίνει στο μέλλον με τις δραστηριότητες μας στη χώρα αυτή. Θα κάνω κάποιες παρατηρήσεις πάνω σε αυτό και πώς εξελίσσονται οι εργασίες αυτές. Καταρχήν να μην ξεχνάμε ότι έχουμε επιτύχει όλοι μας αρκετά μετά το 2002 στη χώρα αυτή, στην εκπαίδευση, την υγεία, και στα, στην καταπολέμηση των ναρκωτικών, τη διακυβέρνηση. Έχει γίνει μεγάλη βελτίωση σε σχέση με το τι γινόταν επί Ταλιμπάν και εμείς πρέπει να ε, πούμε ότι επικεντρωθήκαμε στο νόμο, στο δίκαιο, στη δικαιοσύνη δηλαδή. Ε, δικαιοσύνη ε, κλπ. Ε, ήταν δύσκολες οι αποστολές ε, παρακολούθησης των εκλογών και πρέπει εδώ να καλωσορίσω, να, να συγχαρώ όλους όσους συμμετείχαν και βεβαίως θα συνεχίσω με την παρακολούθηση και στις επόμενες εκλογές. Πάντως, ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο τέλος αυτής της προσπάθειας στο Αφγανιστάν, αλλά μπαίνουμε σε μια τελική φάση ίσως πρέπει να κάνουμε και άλλες προσπάθειες για να βελτιώσουμε την ικανότητα του Αφγανιστάν ε, να, να, βαθμιστεί δηλαδή η διακυβέρνηση σε όλη τη χώρα, να βελτιωθούν οι πολιτικές συμπεριφορές, τις εκλογές, την καταπολέμηση της διαφθοράς, της προστασία δικαιωμάτων γυναικών, παιδιών κλπ. Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να συμβάλλουμε και εμείς σε όλους αυτούς τους τομείς ε, ενισχύοντας τις προσπάθειες της ISAF και άλλων από το στρατιωτικό σκέλος. Σε πρακτικό σημείο θα πρέπει λοιπόν η διαδικασία αυγανοποίησης να συνεχιστεί, ιδιαίτερα ίσως ό,τι αφορά την διοίκηση της χώρας ε, σε υποεθνικό όπως λέμε επίπεδο, σε επαρχίες, στα χωριά, στις πόλεις, ε, όπου αν ξέρετε τη χώρα εκεί είναι τεράστιες οι προκλήσεις. Ιδιαίτερες προσπάθειες θα απαιτηθούν για την εκπαίδευση των αξιωματούχων σε, εθνικό, σε κεντρικό και επαρχιακό επίπεδο. Ε, ε, ε, υπάρχει μια διαδικασία εδώ σε ένα τεράστιο τομέα που πρέπει να βελτιωθούν οι επιδόσεις. Επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παραμείνει σημαντική στην εκπαίδευση αστυνομικών δικαστικών, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν ανθρώπινοι πόροι, οικονομικοί πόροι να διατεθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα στον αστυνομικό τομέα. Συνεργαζόμαστε με την Κομισιόν και ελπίζω και τα κράτη-μέλη να συμβάλλουν. Ε, το δύσκολο θέμα τώρα της ε, επανενσωμάτωσης ε, συμφιλίωσης, εδώ πρέπει να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση ρόλο υποστηρίζοντας το Αφγανιστάν. Θα πρέπει όπου είναι δυνατόν οι εξεγερμένοι να ενσωματωθούν. Όμως το εγχείρημα πρέπει να, στο εγχείρημα πρέπει να ηγούνται οι Αφγανοί. Επίσης η στρατηγική ανάπτυξη του Αφγανιστάν θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το 2013. Νέα όμως μετά το 2010 ε, θα πρέπει να υπάρξει ένα νέο πρόγραμμα. Ε, έχουμε ε, γίνει μάρτυρες κάποια στασιμότητα τώρα. Γι' αυτό οι τελικές συστάσεις της Επιτροπής Εκλογών θα πρέπει να ενσωματωθούν στο μελλοντικό διάλογο στα, στη, σε θέματα διακυβέρνησης και δικαιωμάτων και επίσης θα πρέπει να έχουμε μια στρατηγική μέσων ενημέρωση για να περάσουν οι ιδέες μας. Ε, η Βερονίκα Αρνό θα μας πει περισσότερα για την κατάσταση επιτόπου ε, και με την, αν μου το επιτρέπετε, η κυρία Αρνό θα προσθέσει ορισμένα πράγματα σε σχέση με αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευτυχώς ε, δεν βρίσκομαι σήμερα στο Αφγανιστάν αλλά σήμερα μαζί σας αλλά οργανώσαμε αυτή την επιχείρηση που ήταν αρκετά εξαιρετική. Όπως γνωρίζετε, πρόκειται για ένα σημαντικό πολιτικό μέσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο διευθύνεται από την Επιτροπή που είναι οι παρατηρήσεις στις εκλογές. Έχουμε πείρα εδώ και 20 χρόνια με παρατηρητές των εκλογών, αλλά η επιχείρηση στο Αφγανιστάν ήταν τελείως εξαιρετική. Γιατί, ήδη ότι ήταν οι πρώτες εκλογές εδώ και πολύ χρόνο που, είχαν, ε, που ελέγχονταν και είχαν οργανωθεί από τους Αφγανούς. Το 2005 επίσης είχαμε παρατηρητές, είμαστε και παρόντες το 2004 για να, για να βοηθήσουμε τους Αφγανούς, αλλά εκείνη την εποχή ήταν η διεθνής κοινότητα που ήλεγχε την όλη διαδικασία. Τώρα ήταν η πρώτη φορά που, ε, είχαμε, δοκιμάζαμε τους Αφγανούς για να οργανώσουν εκλογές. Ήταν ε, ιδιαίτερη πρόκληση από την άποψη της ασφάλειας και αυτή η αποστολή είχε εξαιρετικά χαρακτηριστικά στο μέτρο που ε, στείλαμε ανθρώπους ε, δύο μήνες, είχαμε μια ιδιαίτερη υποδομή ασφαλείας και προσπαθήσαμε να έχουμε οκτώ μικρά κέντρα εκτός Καμπούλ, δηλαδή ε, μπορέσαμε να παρακολουθήσουμε τι έγινε στη χώρα κατά τη διάρκεια δύο μηνών, πράγμα που ήταν σημαντικό. Αυτό που ήταν επίσης εξαιρετικό ήταν ότι δεν υπήρχε αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συνήθως αυτό γίνεται, αυτό γίνεται μαζί ή παράλληλα. Ε, έχουμε ε, παρατηρητές μακροπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους και συνήθως έχουμε μια συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με παρατηρητές βραχυπρόθεσμους. Λόγω της κατάστασης στο Αφγανιστάν αυτό δεν κατέστη δυνατόν με την υποστήριξη όλων των κρατών μελών αλλά και του Καναδά, της Νορβηγίας και της Ελβετίας με τις οποίες χώρες έχουμε ειδικέ συμφωνίες και που έχουν πολλές γνώσεις στον τομέα αυτό. Στείλαμε μια μεγάλη ομάδα με περίπου 100 παρατηρητές και όπως σας έλεγα κύριε Πρόεδρε στην Καμπούλ αλλά και σε άλλα 8 περιφερειακά κέντρα με 22 διαφορετικές εθνικότητες συν Καναδούς, Νορβηγούς και Ελβετούς. Ε, η Επίτροπος ε, συνήθως ε, θέλει να έχουμε μια προσωπικότητα κάποιον που να κατευθύνει, να διευθύνει αυτές τις επιχειρήσεις τις εκλογικές, διότι τα πράγματα γίνονται πιο αξιόπιστα από τον αν υπάρχει ένας γραφειοκράτης όπως εγώ ή άλλοι και ακριβώς ένας ευρωβουλευτής έχει ε, μια κατανόηση των εκλογικών μηχανισμών που ίσως άλλοι δεν έχουν. Συνεπώς η Επίτροπος Μπενίτο Φερέρο όταν χρειάστηκε να αποφασίσει πριν από το τέλος της ε, θητείας ε, του παλιού κοινοβουλίου, ζήτησε από τον Φίλιπ Μοριγιόν, ο οποίος ήδη είχε εργαστεί για μας στο Κονγκό και που ε, είχε εργαστεί επίσης στη Βοσνία να αναλάβει αυτή την επιχείρηση που ήταν ιδιαίτερα περίπλοκη και για την οποία νομίζω ότι δεν υπήρχαν δεν υπήρχαν, θα το πω διπλωματικά, δεν υπήρχε πολύς ενθουσιασμός για τις εκλογές στο Αφγανιστάν λόγω των δυσκολιών στον τομέα της πολιτικής και της ασφάλειας. Όσον αφορά στα αποτελέσματα, Δύο μήνες πριν είχαμε παρατηρητές, όπως είπε ο συνάδελφος, ε, διαπιστώσαμε ότι η πλαισίωση νομοθετική η εργασία της Αυγανικής Επιτροπής και της Επιτροπής Παραπώνων Προσφυγών ήταν πολύ καλή εργασία και βρήκαμε ότι στις δύσκολες συνθήκες οργάνωσης αυτών των εκλογών τα πράγματα δεν ήταν τόσο ε, κακά και ότι οι άνθρωποι μετακινήθηκαν πολύ περισσότερο από ό,τι περιμέναμε λόγω των απειλών ε, που είχαν εκφραστεί και που ήταν πραγματικές βεβαίως ε, υπήρχαν, είχαμε πολλούς θανάτους, αλλά μπορέσαμε γενικά να, ε, να, παρακολουθήσουμε ένα μεγάλο μέρος της χώρας, όχι όλη τη χώρα. Επίσης, ε, συνεργαστήκαμε με παρατηρητές τοπικούς ή με παρατηρητές άλλων οργανώσεων που βρίσκονται επί τόπου για να ανταλλάξουμε πληροφορίες. Λόγω των ιδιαιτέρων των ειδικών περιστάσεων, τα πράγματα δεν πήγαν και τόσο άσχημα. Η πλαισίωση νομοθετική και τα δεδομένα δεν ήταν ε, άσχημα, αλλά από την ημέρα των εκλογών κύριε Πρόεδρε, αν κοιτάξετε την προκαταρκτική δήλωση διακήρυξη αναφέρονται ορισμένα προβλήματα τα οποία είναι διαρθρωτικά. Ένα από τα σοβερότερα είναι η έλλειψη ε, εκλογικού καταλόγου ε, που καθιστά τον έλεγχο του αριθμού των ψηφοφόρων και της ποιότητας των ψηφοφόρων πάρα πολύ δύσκολο, κυρίως με ένα ιδιαίτερο πρόβλημα για τις γυναίκες όπως το φαντάζεστε. Άλλα στοιχεία τα οποία ήταν ανησυχητικά ήταν το γεγονός ότι τα μέσα ενημέρωσης έδιναν, ε, ευνοούσαν ε, κάπως ε, τον, τον σημερινό πρόεδρο, αλλά δυστυχώς όπως βλέπουμε σε πάρα πολλές χώρες όπου παρακολουθούμε τις εκλογές αυτό γίνεται και τελικά λέμε ότι το νομοθετικό πάνελ, το πλαίσιο δεν ήταν κακό, αλλά υπάρχουν προβλήματα. Αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι ήμασταν εκεί για να βοηθήσουμε τους Αφγανούς, ήμασταν παρόντες και είμαστε πάντοτε παρόντες. Έχουμε μια σημαντική ομάδα ακόμα και τώρα που βοηθάει και, ε, και βλέπει πώς γίνεται η καταμέτρηση των ψήφων ε, υπάρχουν όλο και περισσότερα θέματα για την οθεία, για αυτό που κάνουμε. Καταγγέλουμε στις αφγανικές αρχές η Επιτροπή των, για τις διαφορές, για τα παράπονα, για τις αιτιάσεις που αποτελείται από πέντε άτομα με τρεις προσωπικότητες που δεν είναι Αφγανοί και αυτό που προσπαθήσαμε να πούμε με τα κράτη-μέλη και την Κομισιόν, είναι ότι κάναμε έκκληση στους υποψήφιους να μην αρχίσουν να θριαμβολογούν και να περιμένουν τα αποτελέσματα. Για την ώρα αυτό έγινε, για την ώρα δεν υπάρχει φίλιος πόλεμος. Οι ε, υποψήφοι μπορούν να ελέγχουν τις ομάδες τους ε, και αναγγέλλονται τα αποτελέσματα βαθμιαία προοδευτικά. Το πρόβλημα που υπάρχει γενικά είναι ότι δεν έχουμε αποτελέσματα για το ποσοστό συμμετοχής όταν ε, βλέπουμε εκλογές εκεί. Πρέπει οι εκλογές να είναι ασφαλείς, να είναι inclusive, να έχουν συμπερίληψη και να είναι αντιπροσωπευτικές. Και το ποσοστό συμμετοχής είναι ένα χαρακτηριστικό σημαντικό. Όλα βεβαίως είναι σχετικά ε, βεβαίως συμμετοχή 40% στην Ευρώπη είναι κάτι το καταπληκτικό. Στο Αφγανιστάν πώς μπορεί κανείς να θεωρήσει ένα 40%. Ένα δεύτερο πράγμα που μας απασχολεί και απασχολεί όλους είναι ότι το γεγονός ότι στο Νότο οι περισσότεροι παρατηρητές τη μέρα των εκλογών δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν καλά τα πράγματα και να παρέμβουν και υπάρχει μια διαφορά συμμετοχής ανάμεσα στο Νότο και στο Βορρά. Και αυτό που είναι προφανές είναι ότι οι συνθήκες ασφαλείας και η απειλή απειλές απέτρεψαν πάρα πολλούς αυγονούς να πάνε να ψηφίσουν και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο ε, θέτει ε, πρόβλημα στο προς, πώς θα θεωρήσουν οι Αυγανοί το αποτέλεσμα. Το γεγονός ότι πολλοί δεν μπόρεσαν να πάνε να ψηφίσουν. Αυτό που παρατηρούμε για την ώρα είναι ότι υπάρχουν υπάρχει περίπου 60% των εκλογικών τμήματων όπου έχει γίνει καταμέτρηση. Ο τρίτος τύπος αποτελεσμάτων που έχουμε, το πρώτο αποτέλεσμα Καρζάη επικεφαλίσα, το δεύτερο είχε μειωθεί, τώρα τα αποτελέσματα σήμερα το πρωί μας δίνουν με 60% των εκλογικών ε, τμήματων, 47,3 ε, για Καρζά, για τον Αμπτουλά Αμπτουλά 30 κάτι, πράγμα που είναι καλό αποτέλεσμα όπως έλεγε ο συνάδελφος και ο τρίτος Μπας Αρντόστα έχει 11,6% αλλά δεν έχουν τελειώσει η καταμέτρηση. Το χρονοδιάγραμμα που έδωσαν οι αρχές του Αφγανιστάν είναι το εξή μα είπαν, είπαν στη διεθνή κοινότητα ότι θα έδιναν προκαταρκτικά αποτελέσματα μεταξύ της 3ης και της 7ης Σεπτεμβρίου. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε στις 3 του μηνός προκαταρκτικά αποτελέσματα, μάλλον προς τις 7 Σεπτεμβρίου προκαταρκτικά αποτελέσματα σημαίνει αποτελέσματα που δεν είναι πιστοποιημένα, διότι εντωμεταξύ υπάρχει το γραφείο των αιτιάσεων, των προσφυγών που θα εξετάσει τις προσφυγές και για την ώρα υπάρχουν πάρα πολλές προσφυγές, 20.000 εκ των οποίων 600 θεωρούνται ότι θα μπορούσαν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα των εκλογών. Θα πρέπει να γίνει κάποια διαλογή, να δούμε πού υπήρξαν ε, συμβάντα, αλλά τα οποία δεν μπορούν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα, αλλά πράγματα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα και όπου θα χρειαστεί ίσως νέα εκλογή. Υπάρχουν ε, λοιπόν σοβαρές αιτιάσεις σημαντικές και είναι μια πρόκληση αυτή. Ε, για την ώρα, ε, όπως είχαν πει 17, θα τελειώσει όλη η δουλειά στις 17 Σεπτεμβρίου. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι ε, τα πιστοποιημένα αποτελέσματα θα μπορέσουν να υπάρξουν μόνο αφού η Επιτροπή των Εκλογικών Προσφυγών θα έχει επικυρώσει τα αποτελέσματα. Αυτό θα γίνει μάλλον στις 17 με ε, ε, αποτελέσματα πιστοποιημένα μεταξύ 17 και 21 Σεπτεμβρίου. Όπως σας είπα κύριε Πρόεδρε, η ομάδα μας είναι πάντοτε παρούσα και προσπαθεί να συλλέξει πληροφορίες και επισύρει τις αρχές πάνω σε κάθε παρατυπία και ανομαλία. Έχουν πρόσβαση στις, ε, στην καταμέτρηση παντού και θα δούμε αν θα γίνει ένας δεύτερος γύρος ή όχι στο Σύνταγμα του Αφγανιστάν προβλέπει ότι υπάρχει δεύτερος γύρος εάν ένας υποψήφιος δεν επιτύχει πάνω από 50% στον πρώτο γύρο. Για την ώρα λοιπόν δεν μπορούμε να πούμε τίποτα και νομίζω ότι αυτά τα οποία είπαμε σε όλους και ενθαρρύνουμε όλους να είναι πάρα πολύ, τους παρακινούμε όλους να είναι πάρα πολύ επιφυλακτικοί και προσεκτικοί διότι με την καταμέτρηση έτσι ως έχει ε, δεν έχουμε τα αποτελέσματα για όλα τα εκλογικά τμήματα και δεν μπορούμε να πούμε ποιος είναι το ποσοστό συμμετοχής, ποια είναι τα αποτελέσματα και ποιες θα είναι οι συνέπειες όλων αυτών των προσφυγών που υπάρχουν. Πρέπει να σας πω ότι ε, οι προσφυγές έχουν γίνει σε όλα τα κόμματα. Ε, θα μου πείτε ότι αυτό δεν είναι καλό αλλά ότι, όλοι παίζουν το παιχνίδι για την ώρα και λένε ότι το σύστημα πρέπει να λειτουργήσει και η εκλογική επιτροπή πρέπει να κάνει τη δουλειά της. Αυτό μπορώ να πω σε αυτό το στάδιο και βέβαια αυτό που θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι οι συστάσεις που η Επιτροπή αυτή, η εκλογική παρατηρητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα κάνει και για να μπορέσουν οι συστάσεις να βελτιώσουν το σύστημα είτε από νομοθετικής απόψεως είτε από πρακτικής και να μπορέσουμε να βελτιώσουμε ακόμα και αν ο χρόνος είναι σύντομος το σύστημα για να μπορέσουμε να ε, βοηθήσουμε την δημοκρατία που οικοδομείται στο Αφγανιστάν, διότι θα υπάρξουν βουλευτικέ εκλογέ τον Ιούνιο του 2010. Δεν έχουμε λοιπόν πάρα πολύ χρόνο μέχρι τότε και θα πρέπει να διορθώσουμε ότι δεν πάει καλά βάσει των συστάσεων των εμπειρογνωμόνων που θα έχουμε μετά τα αποτελέσματα στις αρχές του Οκτωβρίου. Τότε θα έχουμε τις οριστικές συστάσεις των εμπειρογνωμόνων όταν θα έχουμε μια εικόνα της όλης κατάστασης, αλλά σας υπενθυμίζω ότι μας είπαν ότι ήμασταν κάπως αφελείς όταν είπαμε ότι όλα ήταν πολύ καλά. Εμείς δεν το είπαμε αυτό. Είπαμε ότι υπήρχε μια βελτίωση, ότι τα πράγματα ήταν καλύτερα από ό,τι ελπίζαμε στην ε, περιστάσει του Αφγανιστάν. Η κατάσταση δεν είναι όπως στην Νορβηγία και λαμβανομένων υπόψη των συνθήκων ασφαλείας. Είμαστε εκεί για να βοηθήσουμε το Αφγανιστάν να μην δραματοποιούμε τα πράγματα, αλλά να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους βεβαίω και προσπαθούμε να επισύρουμε την προσοχή όλων πάνω στα προβλήματα που διαπιστώσαμε και προσπαθούμε η κανονική διαδικασία εκλογών να τηρηθεί. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαστε στη διάθεσή σας για συμπληρωματικές πληροφορίες. Να ευχαριστήσουμε και τον δόκτορα Μωράν και την δόκτορα Αρνό για την εισήγηση και αρχίζουμε τη συζήτηση. Αρχίζουμε με την επικεφαλής αυτής της πρωτοβουλίας που είναι η κυρία Λούνατσεκ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τους δύο εκπροσώπους της ε, Κομισιόν που πολύ γρήγορα δέχτηκαν να έρθουν και να μας εξηγήσουν τη διεξαγωγή των εκλογών όπως την είδαν και αναφερθήκατε και σε κάποια προβλήματα βέβαια. Ο λόγος ε, για το αίτημα της ομάδας μου να συζητηθεί το θέμα τώρα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έχει Επιτροπή Παρακολούθησης εκεί ακόμα και επένδυσε και πολλά χρήματα. Ε, και κατά τη μέρα των εκλογών και μετά υπήρξε κάποιο πρόβλημα με τις πολύ ενθουσιώδεις παρατηρήσεις σε σχέση με την διεξαγωγή των εκλογών. Γιατί και ο στρατηγός Μοριγιό έλεγε ότι ήταν πολύ καλές, δίκαιες εκλογές και η Επίτροπος Φερέρο Βάλτνερ είπε ότι αποτελούν νίκη για τον ε, αφγανικό λαό και τη δημοκρατία. Και νομίζω ότι αυτός ο ενθουσιασμός ε, κάλυψε, συγκάλυψε κάποια γεγονότα όπως αυτά που είπατε εσείς, ότι δηλαδή υπήρξαν σε μεγάλη κλίμακα προβλήματα. Άρα λοιπόν ήταν λίγο ευσεβής πόθος αυτός ο ενθουσιασμός, αφού φαίνεται ότι υπήρχε η ελπίδα ότι θα ήταν η προσέλευση στις εκλογές μεγάλη, θα συμμετείχε ο πληθυσμός και δεν θέλαμε να δούμε ούτε ως Ευρωπαϊκή Ένωση τα μεγάλα προβλήματα που προέκυψαν και αυτός είναι ένας λόγος ε, που θέλαμε να συζητηθεί το θέμα. Τα πάτε κι εσείς εν μέρη. Υπήρξαν επικρίσεις, υπήρξαν περίπου 3.000 ε, προσφυγές ε, στην Επιτροπή Προσφυγών στις εκλογές για πλέον πλέον διαφορετικούς λόγους, ότι τα ψηφοδέλτια ήταν λάθος, ότι ήταν περισσότερα από αυτά που έπρεπε, ότι χάθηκαν κάποιες κάλπες ότι ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις γυναίκες ε, ε, πήγαν κάποιοι να ψηφίσουν για λογαριασμό των γυναικών και δεν πήγαν οι ίδιες και αυτό το Ίδρυμα για το Free and Fair Elections είπε ότι 650 εκλογικά τμήματα, ειδικά για τις γυναίκες, είχαν κλείσει, δεν ήταν ανοιχτά κατά την ημέρα των εκλογών και 1050 ε, εκλογικά τμήματα τη μέρα των εκλογών άνοιξαν μία ώρα μετά την ε, συγκεκριμένη ώρα. Επίσης υπήρξαν πολλές απειλές από τις κυβερνητικές αρχές και τοπικές αρχές. Ε, κάποιους ισχυρούς άντρες δηλαδή σε τοπικό επίπεδο που επέβαλαν ποιος έπρεπε να ψηφιστεί. Όλα αυτά λοιπόν δεν ήταν free and fair, ελεύθερες και δίκαιες εκλογές και επίσης ε, πήγαν να ψηφίσουν περισσότεροι από αυτούς που φοβόμαστε αρχικά. Στο Νότο όμως δεν συνέβη αυτό καθόλου. Δεν πήγαν. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι ότι οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θεώρησαν ότι όλα πήγαν θαυμάσια. Το, το υπερβάλλω λίγο τώρα αυτό που λέω. Εν πάση περιπτώσει, στην πραγματικότητα δεν έγιναν έτσι. Αντίθετα, υπήρχε τεράστιο πρόβλημα. Γιατί δεν έπρεπε να γίνουν αυτά. Ε, τώρα θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ποιες δυσκολίες υπήρξαν, θα πρέπει να διευκρινιστεί σε ποιο βαθμό ε, πρόκειται για εκλογική απάτη ή νοθεία και από το αποτέλεσμα θα πρέπει να ξεκαθαρίζεται το θέμα. Πήρε όντως, έχει όντως την πλειοψηφία ο ή όχι. Γιατί Ίσως θα πρέπει να υπάρξει ένα δεύτερο γύρο για να διευκρινιστεί το θέμα. Ο Αμπτουλά Αμπτουλάη είπε ότι είδε και εκείνο κάποιες ε, τέτοιου είδους ε, νοθείες. Ε, ένας Γερμανός στο Αφγανιστάν που είχε εργαστεί για το ίδρυμα αυτό στο Βερολίνο εδώ και πολλά χρόνια και είχε συμμετέχει στην αποστολή των Ηνωμένων Εθνών για το στο Αφγανιστάν, λέει και παραθέτω τώρα ότι και για αφγανικά δεδομένα οι εκλογές δεν ήταν πολύ καλές. Και η γνώμη του είναι ότι πρέπει να υποθέσουμε ότι υπήρξε εκλογική νοθεία, ξέρει το Αφγανιστάν εδώ και χρόνια, γνωρίζει την κατάσταση και είναι γι' αυτό βαρύνουσες αυτές οι απόψεις. Γι' αυτό ήταν λίγο ενοχλητικό το γεγονός ότι από πλευράς Ευρωπαϊκή Ένωση όλα αυτά δεν λήφθησαν σοβαρά υπόψη. Ε, δεν μπορούμε δηλαδή να ευχόμεθα απλώ, να εκφράζουμε ευχέ και να λέμε όλα πάνε πολύ καλά στο Αφγανιστάν, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι. Θα περίμενα μεγαλύτερη προσοχή από την Κομισιόν και την Επίτροπο. Ξεκάθαρα λόγια να πούνε δηλαδή ότι τόσο καλά δεν ήταν τα πράγματα όπως είπαμε στην αρχή. Αυτό θα βοηθήσει και τη χώρα και το λαό του Αφγανιστάν που περιμένει να δει πού θα οδηγήσουν όλα αυτά. Να ξεκαθαριστεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση που είχε εκπροσώπηση εκεί και που είναι συνδεδεμένη με πολλές ελπίδες από το λαό αυτών, η Ευρωπαϊκή αυτή Ένωση δεν παραγνωρίζει τα ε, πραγματικά και υφιστάμενα προβλήματα. Αυτό είναι μια ε, οφειλή που έχουμε και προς τον εαυτό μας και προς το λαό του Αφγανιστάν. Γι' αυτό λοιπόν ε, ε ήθελα να κάνω τις ερωτήσεις μου. Μας είπατε για τα προσωρινά εκλογικά αποτελέσματα. Θα με ενδιαφέρει επίσης να μάθω την εκτίμησή σας ε, της κατάστασης ε, και των σχέσεων Αμπτουλά, Καρζάη Αμπτουλά είπατε ότι δεν, ε, υπήρξαν, δεν σημειώθηκαν έκτροπα, ευτυχώς. Τώρα περιμένει ο κόσμος να δει ποια θα είναι τα αποτελέσματα, αλλά θα με ενδιέφερε η δικιά σας η εκτίμηση. Δηλαδή, όταν θα κοινοποιηθούν τα αποτελέσματα, τι αντιδράσεις θα υπάρξουν. Ας πούμε, 55% κέρδισε ο Καρζάη. Αν βγει αυτό το αποτέλεσμα, αν ο Αμπτούλα Αμπτούλα πάρει το 40%. Ε, είναι ε, περίεργα τα αποτελέσματα, μικρές διαφορές. Τι θα γίνει στο μέλλον. Ενδέχεται να συνεργαστούν στο μέλλον οι δύο αυτοί άνδρες. Τι πληροφορίες έχετε απευθείας άμεσα από το Αφγανιστάν. Ε, αυτά μας ενδιαφέρουν να τα μάθουμε. Και όπως σας είπα υπάρχει αυτή η κριτική ότι στην αρχή και στη, από τις δηλώσεις ε, και της Επιτρόπου και του κυρίου Μοριγιόν ε, φάνηκε ότι περισσότερο ευσεβείς πόθους εκφράζουμε παρά ε, αντικατοπτρίζομαι και δείχνομαι ε, μια εμπεριστατωμένη ανάλυση των γεγονότων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αλαφράνκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εκπρόσωπο της Επιτροπής. Ευχαριστώ που απαντήσατε τόσο σύντομα στην πρωτοβουλία μας, την κοινοβουλευτική. Θα ήθελα να σας πω εξ αρχής ότι δεν συμφωνώ με τους ισχυρισμούς της συναδέλφου την υποστήριξα στο αίτημά της, ούτως ώστε η Επιτροπή να μοιραστεί μαζί μας της πληροφορίας. Η ε, αποστολή παρατηρητών ε, για τις εκλογές είναι κάτι το ουσιαστικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πρόκειται για αποστολές που είναι ανεξάρτητες. Είπατε ότι όντως ίσως υπερβάλλατε σχετικά με τον ενθουσιασμό στις δηλώσεις της Φερέρο Βάλτνερ σε αυτά τα οποία είπε ο στρατηγός Μοριγιό, αλλά εγώ διάβασα τα όσα είπε η Επίτροπος Φερέρο Βάλτνερ. Ε, είδα αυτή την δήλωση του στρατηγού Μοριγιό και νομίζω ότι το μόνο πράγμα που μπορούμε να πούμε ότι δεν βλέπουμε κανέναν ενθουσιασμό διότι στην πρώτη παράγραφο ε, της ε, δηλώσεως της ε, Επιτρόπου βλέπουμε μια επιδείνωση της κατάστασης και ο στρατηγός Μεριγιόν λέει ότι υπάρχουν 11 άτομα τα οποία πέθαναν, υπήρξε μια απόπειρα με, ε, με βόμβα σε αυτοκίνητο με 40 νεκρούς, είδαμε τι συνέβη στα μέσα ενημέρωσης ότι κόψανε στο ανθρώπου στο χέρι ή τη μύτη επειδή συμμετείχανε στις εκλογές. Δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει πραγματικός ενθουσιασμός. Μιλάμε εδώ για προκαταρκτικές δηλώσεις, αλλά ότι μιλάμε για προκαταρκτικά ξέρουμε τι εννοεί αυτό και πώς λειτουργεί λειτουργούν οι αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει ε, να δούμε την εκλογική διαδικασία στο σύνολό της και αυτό πρέπει να γίνει μέσα τρεις μέρες μετά τις εκλογές. Αλλά το ξέρετε καλά αγαπητοί συνάδελφοι, αυτή η διαδικασία η εκλογική δεν μπορεί να εστιαστεί μόνο στην ημέρα των εκλογών. Πρέπει να μιλήσουμε για το σύνολο της διαδικασίας, πώς λειτουργήσε η εκλογική επιτροπή, αν ήταν ανεξάρτητη, αν ήταν μια διοίκηση που μπόρεσε να διευθετήσει ορισμένες διαφορές, αν κάθε υποψήφιος μπόρεσε να εκφραστεί στα μέσα ενημέρωσης, αν όλη η διαδικασία ήταν ε, δίκαιη. Ξέρουμε ότι υπήρξαν προβλήματα στην διαδικασία την εκλογική. Ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση στο Αφγανιστάν. Κύριε Πρόεδρε, εγώ προείδρευσα μια αποστολής εκλογική σε αυτή τη χώρα. Ήμουν πρόεδρος, ήταν και επίση ο στρατηγός μοριγιών τότε. Νομίζω ότι πάρα πολύ λίγοι συνάδελφοι μπορούν να πούν ότι έχουν τόση πείρα, ε, τόση τεχνογνωσία όσο ο, ο στρατηγός Μοριγιό εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να υποστηρίξουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έκανε τα όσα έκανε. Βεβαίως αυτές οι αποστολές κοστίζουν πολλά χρήματα, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση κοστίζουν χρήματα για το σύνολο της διεθνούς κοινότητας, αλλά πρέπει να ενισχύσουμε αυτήν την δημοκρατική πρωτοβουλία. Αλλά αυτά πρέπει να τα κηρύσουμε, αλλά θα πρέπει επίσης να δράσουμε, να είμαστε πρωταγωνιστές για να αγωνιστούμε για την ειρήνη, για τον εκδημοκρατισμό, για την υπόθεση της ειρήνης στη χώρα αυτή. Αυτά, αυτά. Θα έλεγα λοιπόν ότι από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδείξαμε πολύ θάρρο, στείλαμε μια τεχνική αποστολή επιτόπου, προσπαθήσαμε να διευκολύνουμε αυτήν την αποστολή ε, εκλογικών παρατηρητών και είχαμε τον στρατηγό Μοριό, ο οποίος ήταν το καταλληλότερο πρόσωπο για να πάει επί τόπου. Όλα λοιπόν τα όσα είπατε, ε, δεν ξέρω. Εγώ διάβασα τις δηλώσεις της Επιτρόπου, διάβασα τις ε, δηλώσεις του στρατηγού Μοριγιό και δεν ε, συμφωνώ με τα όσα είπατε εσείς. Αυτό το οποίο εμείς πρέπει να κάνουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να υποστηρίξουμε τους εκπροσώπους μας. Θα πρέπει τώρα ε, να είμαστε υπομονετικοί και να δούμε πώς θα επιλύσουμε αυτές τις περιπτώσεις νοθείας. Υπήρξαν πολλές νοθείες, αλλά έχουμε εδώ όργανα τα οποία μπορούν να δράσουν όπως και θα πρέπει. Και θα πρέπει να αποφύγουμε, να βιαζόμαστε, να εξαγάγουμε συμπεράσματα. Ίσως να υπάρξει ένας δεύτερος γύρος. Μην ξεχνάτε ότι έλαβαν χώρα οι εκλογές σε μια πολύ τεταμένη δραματική κατάσταση. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να συγχαρούμε τον αφγανικό λαό, ο οποίος απήντησε μαζικά σε αυτήν την έκκληση, ε, σε αυτό το κάλεσμα για να ψηφίσει. Ας περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα να έχουμε οριστικά αποτελέσματα και όχι προσωρινά. Το όργανο το οποίο θα ασχοληθεί με τις προσφυγές θα μπορεί να μας πει αν υπήρξαν, υπήρξε νοθεία νοθεία σημαντική για να μπορέσει να τεθεί ένα αμφιβόλο, να αμφισβητηθεί όλη η εκλογική διαδικασία. Ενώ αυτό το όργανο δεν θα έχει αποφασίσει, εμείς θα πρέπει να βοηθήσουμε, να συγχαρούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έδρασε εξαίρετα, που διευκόλυνε αυτήν την αποστολή των παρατηρητών και θα πρέπει τον πρώην συναδελφό μας, τον στρατηγό Μοριό, να τον συγχαρούμε διότι εργάστηκε πολύ για αυτή την υπόθεση που είναι κοινή μας υπόθεση, υπόθεση του Κοινοβουλίου μας. Ευχαριστούμε τον κύριο Σαλαφράγκα. Ο κύριος Ομπιόλς έχει το λόγο. Τι είναι αυτό? Πρόεδρε, ο ειδικό εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Αφγανιστάν και Πακιστάν δυστυχώς δεν βρέθηκε εδώ μαζί μας και θα ήθελα να πω ότι η παρουσία του μαζί με τον φίλο μας, τον κύριο Μοριγιόν, θα οδηγούσε σε μια συζήτηση όχι μόνο σε σχέση με τη διενέργεια των εκλογών στο Αφγανιστάν, αλλά και με τη γενικότερη κατάσταση. Νομίζω Ε, ε, ε, από όσο γνωρίζω κάποιος αναφέρθηκε στο ότι ένας από τους στόχους είναι να υπάρξει συνοχή των φυλών της Ευρώπης έναντι εκείνων του Αφγανιστάν. Αυτό λέχθη. Και θα ήθελα να κάνω μια έκκληση στις ευρωπαϊκές φυλές μέσα σε εισαγωγικά, έτσι ώστε να έχουμε ενία φωνή. Πρόκειται για την κλασική συζήτηση για το κατά πόσο ένα ποτήρι είναι μισοάδιο ή μισογεμάτο. Μπορούμε λοιπόν να ε, συμπέσουμε, να προβούμε σε μία ε, σύγκληση απόψεων, δηλαδή η διενέργεια των εκλογών ε, είναι πολύ θετική και αντικατοπτρίζει την τραγική κατάσταση του Αφγανιστάν. Θα πρέπει όμως να μην ε, ακολουθούμε μία πολιτική για την πολιτική. Νομίζω ότι η συζήτηση αυτή εκρεμεί στο Κοινοβούλιο τη στιγμή που στις ΗΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι κυβερνήσεις μιλούν για την κατάσταση του Αφγανιστάν σε μία κρίσιμη καμπή. Ο κύριος Μόραν μίλησε για την επέκταση δυνάμεων στο Αφγανιστάν. Δεν πρέπει να ξεχνά ότι η μεγαλύτερη δύναμη είναι η δύναμη των Ταλιμπάν και άρα θα πρέπει να προβούμε σε μία εις βάθος συζήτηση για το πώς να ανταποκριθούμε σε αυτή την δραματική κατάσταση. Εκρεμεί αυτή η συζήτηση, δεν μπορεί να γίνει σήμερα, όμως ε, νομίζω κύριε Πρόεδρε ότι θα έπρεπε ο κύριος ε, Έτορε Σέκη και ο κύριος Μοριγιόν να βρεθούν εδώ μαζί μας πριν ε, ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση για να είμαστε και σοβαροί. Ευχαριστούμε κύριε Ομπιόλς. Ο κύριος Μέγερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πράγματι ε, δέχομαι την τελευταία παρέμβαση. Θα πρέπει να ε, γίνει μία εις βάθος συζήτηση η ενωτική αριστερά είδα από το 2001 δεν συμμερίστηκε την ε, στρατιωτική εισβολή στο Αφγανιστάν. Ούτε την υποστηρίζουμε τώρα γιατί πιστεύω ότι θα πρέπει να σταματήσει αυτή η φεουδαρχία ιδιαίτερα ως προς τη θέση της γυναίκας καθώς και η παραγωγή οποίου. Δεν δεχόμαστε αυτή την κατάσταση αλλά ούτε την στρατιωτική εισβολή. Αυτές οι εκλογές γίνονται για, εσωτερική, για την εσωτερική κατανάλωση των χωρών που ε, προώθησαν την στρατιωτική εισβολή. Δεν δεχόμαστε λοιπόν την θέση αυτή και θεωρούμε ότι έχει αποτύχει αυτή η στρατηγική. Εμείς ε, θεωρούμε ότι η πραγματικότητα είναι άλλη. Έχουμε δύο υποψηφίους, τον Καρσάη και τον Απτουλάχ. Ο Απτουλάχ δεν είναι τόσο ε, ζηλωτής όπως ο Καρζάη, γιατί όπως ξέρετε ο Καρζάη πρόθυσε νόμους για την γυναίκα που ανήκει στους Σιήτες. Και η θέση της Αφγανής γυναίκας είναι απαράμιλη, ίδια και απαράλλακτη από το 2001 και οι γυναίκες δεν ψήφισαν. Οι περισσότερες γυναίκες ζουν αυτή την φρίκη. Ε, ζουν σε κατάσταση συνεχούς χρήσης της ε, μπούρκας και θεωρούμε ότι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη διότι ο Αύγουστος ήταν ο χειρότερος μήνας. Μόνο οι ΙΠΑ χάσανε 47 στρατιώτες. Χτες ε, πέθανε, σκοτώθηκε ο υπαριθμόν 2 της ΚΥΠ του Αφγανιστάν. Καθώς, και, καθώς μας είχε πει και η κυρία Μαλαλάη Χόγια εδώ και δεν μπορεί να ζήσει ελεύθερα. Πρέπει να ζει σε κατάσταση, πρέπει να ζει σε ένα κρυσφύγετο. Θα πρέπει λοιπόν να δοθούν απαντήσεις ουσίας, διότι σε μία τέτοια κατάσταση πολέμου δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι διενεργήθηκαν ελεύθερες και δημοκρατικές εκλογές δεν πρέπει να εμένουμε ε, στις δικές μας αξίες, δηλαδή ότι οι μορφές διακυβέρνησης πρέπει να ακολουθούν τα δικά μας πρότυπα. Μπορεί να υπάρχει καλύτερη διακυβέρνηση και με άλλους τρόπους. Ε, βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή και θα πρέπει να προωθήσουμε μια ουσιώδη συζήτηση, ουσιαστική συζήτηση Δηλαδή είτε ε, κερδίσει ο Αμπτουλάχ είτε ο Καρζάι, ε, κερδίζουν οι πολεμοχαρείς, οι άρχοντες του τρόμου, όχι οι γυναίκες. Γι' αυτό δεν μπορούμε να τασόμαστε υπέρ της ε, στρατιωτικής παρουσίας. Θα πρέπει να αλλάξουμε την στρατηγική τον ΗΠΑ που είναι μια στρατηγική πολέμου, καθαρή στρατηγική πολέμου, έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ήθελε την εθνική ανοικοδόμηση της χώρας. Αυτή είναι η θέση της ομάδας μου. Δέχομαι αυτά που είπε και ο κύριος Ομπιόλς. Θα πρέπει να προωθήσουμε μια συζήτηση ουσίας μετά από 8 χρόνια στρατιωτικής παρουσίας και εισβολής. Δεν θα πρέπει να ε, ακολουθήσουμε μια διαφορετική στρατηγική επιτέλους. Ευχαριστούμε τον κύριο Μέγερ. Ε, ο κύριος Άτκινς έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πολλά από αυτά που ήθελα να πω έχουν λεχθεί. Συμφωνώ με τη συνάδελφο Λούνατσεκ σχετικά με τη γενική προσέγγιση. Προσυπογράφω κάποιες παρατηρήσεις που έγιναν σχετικά με το αμφίβολο αποτέλεσμα και υπάρχει κάποια αμέλεια εδώ σε σχέση με την ανάλυση γιατί και οι δημοσιογράφοι και άλλοι παρόντες δείχνουν ότι Περίπου 2.500 προσφυγές έχουν γίνει όλων των ειδών ε, και αφορούν και το προσωπικό που εργάστηκε εκεί στα εκλογικά τμήματα και ο κύριος Χολμπουρούκ είχε μια σκληρή συνάντηση με τον πιθανό νικητή και πιστεύουν και εκείνοι ότι πρέπει να γίνει νέος γύρος εκλογών Υπάρχει μεταξύ Παστούν και του λοιπού Αφγανιστάν ε, μία ε, διέρεση που τη δείχνουν οι δύο υποψήφοι και ο ιτημένος δεν θα δεχτεί αν υπάρχει απάτη το εκλογικό αποτέλεσμα και οι υποστηρικτές του θα, κάνουν, και εκείνοι θα τον μιμηθούν. Ε, ελπίζω να προλάβω να πάρω την απάντηση γιατί πρέπει να προλάβω την πτήση μου. Πάντως, η Κομισιόν δεν συμφωνεί ότι ο κύριο Χόλμπρουκ, ένα ε, σεβαστό Αμερικανός και διπλωμάτη ε, όταν εκείνο λέει ότι πρέπει να ξαναγίνουν εκλογές, δεν πρέπει να συμφωνήσουμε κι εμεί. Επίσης, υπάρχει κάποια ένδειξη ότι το αποτέλεσμα των ε, συμβάσεων που έχουν ε, δοθεί από την αφγανική κυβέρνηση ή τους υποστηρικτές που δίνονται ως επιτοπλίστων, ανατίθενται δηλαδή ε, σε εξωτερικούς, εξωτερικ, επιχειρήσεις του εξωτερικού, δεν επηρεάζει τους Αφγανούς που πιστεύουν ότι δεν συμμετέχουν ε, ισότιμα. Επίσης, ποιες ε, ενδείξεις υπάρχουν πριν, κατά τη διάρκεια, μετά τις εκλογές ή και στο μέλλον γενικά ότι το Πακιστάν μπορεί να κλείσει τα σύνορα με δεδομένο ότι ε, ένα σημαντικός αριθμός των ταραξιών έχουν την έδρα τους μάλλον στο Πακιστάν και όχι στο Αφγανιστάν. Πρέπει λοιπόν και αυτό το θέμα να ε, το δούμε ως θέμα ε, προτεραιότητας διπλωματικής, στρατιωτικής αλλά και κοινή λογικής. Επίσης ένας αριθμός Βρετανών στρατιωτών έχασαν τη ζωή τους εκεί και όπως και, από και άλλοι στρατιώτες από άλλα κράτη και είναι δύσκολο να δικαιολογήσουμε την ε, παρουσία μας εκεί. Είναι δύσκολο να δικαιολογήσουμε στους συγγενείς ε, στρατιώτη που πέθανε στο Αφγανιστάν, που σκοτώθηκε στο Αφγανιστάν, ε, να δικαιολογήσουμε ότι οι εκλογές αυτές γίνονται για την επίτευξη δημοκρατικού σκοπού. Να πούμε δηλαδή στα, στις οικογένειες των θυμάτων ότι κάποιοι στρατιώτες σκοτώθηκαν υπερασπιζόμενοι ένα εκλογικό τμήμα όπου μόνο τρεις άνθρωποι μπόρεσαν να πάνε να ψηφίσουν. Είναι πολύ δύσκολο να ε, δικαιολογήσουμε μια τέτοια κατάσταση που αποδεικνύει ότι δεν έχουμε κάνει ότι είναι δυνατόν για να λυθεί το πρόβλημα. Δεν μπορούμε να παίρνουμε λοιπόν ημίμετρα. Πρέπει να φροντίσουμε ε, ολόψυχα το ζήτημα αυτό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πλεύρης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω κάποια σκέψη και εγώ να προσθέσω σε αυτά τα οποία υπόθηκαν. Θεωρώ κύριοι συνάδελφοι ότι κάνουμε μια συζήτηση για τις εκλογές στο Αφγανιστάν, όμως τόσο η διεθνής κοινότητα όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν στυλίτευσε στο βαθμό που θα έπρεπε ότι λίγο πριν τις εκλογές υπήρξε ένας νόμος, η εφαρμογή ενός νόμου κατά των γυναικών που ουσιαστικά προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Και από εκεί και πέρα όταν έχουμε να κάνουμε για μια, ε, ένα τέτοιο περίγραμμα όπου ουσιαστικά η γυναίκα αντιμετωπίζεται ως πράγμα, ως αντικείμενο και από την άλλη πλευρά έχει το δικαίωμα να ψηφίζει, αλλά εφαρμόζονται εις βάρος της όλοι αυτοί οι νόμοι, μπορούμε να καταλάβουμε ότι σε μεγάλο βαθμό όσο και να θέλουν κάποιοι να παρουσιάσουν μια εικόνα ότι υπήρξε μια δημοκρατική επίφαση στις εκλογές του Αφγανιστάν, το Αφγανιστάν είναι πολύ μακριά από αυτό το δρόμο. Δεν έχουμε βέβαια την απέτηση εδώ πέρα το Αφγανιστάν να είχε εκλογές όπως θα είχαν οι ευρωπαϊκές χώρες, αλλά από την άλλη πλευρά δεν είναι δυνατόν είτε από πιέσεις που προέρχονται από τις ΗΠΑ, Αμερικής, είτε από πολιτικές προτιμήσεις που υπάρχουν, να μην βλέπουμε την πραγματικότητα. Θα κλείσουν 10 μέρες περίπου εκλογές στο Αφγανιστάν, δεν θα έχουμε τα αποτελέσματα. Καταγγελίες για νοθεία υπάρχουν παντού. Ε, πολλοί κόσμος δεν μπόρεσαν να πάει να ψηφίσει απορώ πώς μέσα σε όλο αυτό το περίγραμμα μπορούμε να πούμε ότι υπήρξαν κάποια θετικά στοιχεία ώστε να είμαστε αισιόδοξοι για την πορεία. Πράγματι η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένας ε, παράγοντας σε όλη αυτή την περιοχή πρέπει να έχει ένα ενδιαφέρον και πρέπει να έχει ενδιαφέρον και στην κατεύθυνση της ε, θεμελίωσης δημοκρατικών αρχών και την ε, ουσιαστικά κατοχήρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως παράλληλα δεν πρέπει να ξεχνάμε και λόγω αυτής όλης της κατάστασης που έχει προκληθεί, έχουμε μια τεράστια μεταναστευτική ροή από αυτήν τη χώρα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια μεταναστευτική ροή που μπορεί να την πληρώνουν αυτή τη στιγμή πρωτίστως οι μεσογειακές χώρες. Αν όμως δεν ληφθούν μέτρα για να επιστρέψουν αυτοί οι άνθρωποι πίσω και να μπορέσουν εκεί πέρα στη χώρα τους να ζήσουν, είναι βέβαιο ότι στην πορεία θα το πληρώσει και ολόκληρη η Ευρώπη. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να ρωτήσω εάν τυχόν πιστεύουν ότι κάτω από τις συνθήκες στις οποίες έγιναν οι εκλογές τελικά μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ένα αποτέλεσμα που εκφράζει τη βούληση του λαού του Αφγανιστάν. Ευχαριστούμε τον κύριο Πλεύρη. Ο κύριος Σατάρτ Μοντάλτο το έχει το λόγο. Ε, ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα μιλήσω αγγλικά. Ε, ο τρόπος που εξελίσσεται η συζήτησή μου δίνει την εντύπωση ότι ορισμένα μέλη δεν γνωρίζουν καλά την πραγματική σημερινή κατάσταση στο Αφγανιστάν, επιτόπου. Εάν κάποιος περίμενε ε, μια φυσιολογική εκλογή στο Αφγανιστάν, ε, τότε αυτός είναι αφελής. Δεν είναι θέμα ε, του, ανάμεσα να έχει κανείς ελεύθερες και δίκαιες εκλογές. Εκεί το θέμα που ετίθετο ήταν να, γίνουν εκλογές ή να μην γίνουν. Η κατάσταση επιτόπου είναι πολύ χειρότερη από ό,τι φαντάζεται κανείς. Όταν ήμουν στο Αφγανιστάν, ήμουν πρώην μέλος ε, μιας ειδική επιτροπής σχέσεων με το Αφγανιστάν και εκεί καταλαβαίνει κανείς ότι υπάρχει κάποια μορφή διακυβέρνησης, μόνο κάποια μορφή διακυβέρνησης ε, στις αστικές περιοχές και σε ορισμένα τμήματα. Η υπόλοιπη χώρα ε, δεν κυβερνάται ουσιαστικά. Η υπόλοιπη χώρα ζει με τρόμο, η ασφάλεια είναι κάτι το εκτός τόπου και ε, ε, είναι δύσκολο να υπάρχουν εκλογές σε μια εμπόλεμη ζώνη. Προσπαθούμε να έχουμε, νομίζω, σε αυτή τη συζήτηση, ορισμένες παραμέτρους που δεν μπορούν όμως να εφαρμοστούν, να ισχύσουν για το Αφγανιστάν, διότι όλοι γνωρίζουν ότι πρόκειται για μια ειδική περίπτωση η οποία δεν μπορεί να ακολουθήσει τους κοινού κανόνες. Ε, δεν υπάρχουν αναλογίες αλλού. Υπάρχει ένας πόλεμος εκεί που μένετε και δεν είναι ε, ε, θέμα του αν θα ενθαρρυνθούν οι άνθρωποι να ψηφίσουν ή το αντίθετο. Απειλούνται για να μην ψηφίσουν. Και εάν προσπαθούμε να δούμε αν αυτές, αν αυτές οι εκλογές ήταν τελικά επιτυχημένες ή όχι, τότε θα πρέπει όλοι μας να παραδεχθούμε ότι δεν ήταν πιθανόν ελεύθερες, δεν ήταν πιθανόν δίκες, διότι δεν μπορεί κανείς να έχει εκλογές σε μια χώρα που στο εσωτερικό της έχει πόλεμο. Αλλά ποια είναι η εναλλακτική λύση. Η εναλλακτική λύση θα ήταν να μην υπάρξουν καθόλου εκλογές δεν υπήρχε εναλλακτική λέση. Είτε να υπάρξουν εκλογές είτε να μην υπάρχουν. Δεν είναι θέμα του ανεπρόκειτο να υπάρχουν ε, τρομερές εκλογές ε, με φυσιολογικές συνθήκες. Οι συνθήκες δεν είναι καθόλου φυσιολογικές. Όταν ήμασταν ε, στο Αφγανιστάν έτσι ήταν τα... νομίζετε ότι η Καμπούλ είναι ασφαλής, αν το πιστεύσετε, ξεχάσετε το. Δεν μπορεί κανείς να βγει από το ξενοδοχείο του, να περπατήσει στο δρόμο εκτός αν είναι απλισμένος Και με αυτές τις περιστάσεις νομίζω ότι το να μην υπήρχαν εκλογές θα είχε τελικά δείξει ότι όλες οι προσπάθειες που καταβάλλονται για να υπάρξει κάποια ε, μορφή φυσιολογικής ζωή στο Αφγανιστάν θα είχαν αποτύχει. Είναι ωραία να μιλάμε για τις ε, οι γυναίκες, ε, για τις ε, γυναίκες οι οποίες φοράνε την μπουρκα και οι οποίες γυρίζουν πίσω στο 2000 αλλά η κατάσταση που υπάρχει στο Αφγανιστάν και ήμουν παρόν με τον στρατηγό για αρκετό χρόνο εκεί είναι μια κατάσταση όπου αν δεν ελάμβαναν χώρα εκλογές νομίζω ότι ο σκοπός όλης της προσπάθειας που καταβάλλεται από τον ελεύθερο κόσμο ε, σχετικά με το Αφγανιστάν θα είχε πλήρως απαξιωθεί. Ευχαριστώ πολύ. Τέλος, η κυρία Νέιτς έχει το λόγο. Uh, President, your colleagues. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Δεν είμαι μια ειδική του Αφγανιστάν. Ο κύριος Μοριγιό ήταν ο ειδικό της ομάδας μας και ο οποίος ήταν επικεφαλής αυτής της αποστολής παρατήρησης των εκλογών. Αυτό το οποίο θα ήθελα να προσθέσω σχετικά με τις ευρύτερες προσπάθειες παρατήρησης εκλογών και είχα την τιμή να διευθύνω μια ομάδα με συνθήκες που ήταν ε, ε, παραδυσένεια σε σχέση με το Αφγανιστάν ήταν στη Ζάμπια πριν από μερικά χρόνια είναι ότι κάποιος πρέπει να συνειδητοποιεί την πίεση, την πίεση για να υπάρξει μια δήλωση ακριβώς μετά ε, το κλείσιμο των εκλογικών τμήματων. Δεν μπορεί κανείς να καθυστερεί μια δήλωση για μέρες και μέρες και μέρες. Πρέπει λοιπόν μέσα σε δύο-τρεις μέρες να υπάρξει μια δήλωση και αυτό είναι πάντοτε μια δύσκολη πράξη εξισορροπητική. Και είναι δύσκολο εξ αποστάσεως να πει κανείς τι έπρεπε να γίνει, ίσως δεν έπρεπε να πω το ένα ή το άλλο, ότι ο αφγανικός ε, λαός ε, ψήφισε μαζικά ότι είναι μια ε, νίκη για την δημοκρατία, διότι αυτό μπορεί να παρερμηνευτεί, αλλά ζητώ κάποια κατανόηση για αυτή την πίεση, διότι γενικά δεν ξέρω αν αυτή ήταν η περίπτωση στο Αφγανιστάν επίσης, οι αποστολές παρατήρησης Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι οι μόνες επιτόπου συνήθως. Και όσο καν κανείς προσπαθεί να έχει αρμονία με τις άλλες αποστολές, υπάρχει κάποια στιγμή όπου κάτι πρέπει να λεχθεί και προσπαθεί ο καθένας να βρει ένα κοινό μήνυμα με τρόπο ισορροπημένο. Θα ζητούσα λοιπόν περισσότερη κατανόηση για τις διατυπώσεις και τη φρασιολογία που χρησιμοποιήθηκε. Ελέγχθηκε από τους δύο εκπροσώπους της Επιτροπής, όπως είπα και κάποτε στη Ζάμπια, μέχρι, δεν έχουν, μέχρι να έχει καταμετρηθεί και η τελευταία ψήφος δεν θα έχουν τελειώσει τα πράγματα. Και σε περιστάσεις τόσο δύσκολες όπως αυτές του Αφγανιστάν, ε, και με τις ε, καθυστερήσεις, μεγάλες καθυστερήσεις για τον υπολογισμό, η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη. Ακόμη και αν έχω μια αυθόρμητη, ένα αυθόρματο θαυμασμό θα έλεγα για τον κύριο Χάουλμπρουκ. Δεν νομίζω ότι ήρθε ο χρόνος να δηλώσουμε ε, δημόσια ότι ένας δεύτερος γύρος είναι επιθυμητός, είναι πολύ νωρίς. Ποιοι είμαστε εμείς για να πούμε κάτι από, βλέποντας τα πράγματα απ' έξω. Εάν οι Αμερικανοί για κάτι εκλογές σε μια χώρα από τις δικές μας λένε όλα είναι καλά, αλλά θέλουμε να έχετε δεύτερο γύρο». Βεβαίως, ε, αν η διαφορά είναι μικρή ανάμεσα στους δύο υποψήφιους. Αν γινόταν σε εμά θα εξοργιζόμασταν. Είναι δύσκολα τα πράγματα, είναι πολύ λεπτά. Θα ήθελα να συγχαρώ όλη την αποστολή ε, για την εργασία που έκανε με δύσκολες περιστάσεις, αλλά βεβαίως η δουλειά αυτή δεν τελείωσε. Αυτό είχα να πω το πρώτο. Το δεύτερο, θα ήθελα να υποστηρίξω την πρόταση που κάνατε εσείς κύριε ε, και εσείς. Πιστεύω ότι είσαστε και νομίζω και ότι η εκπρόσωπος για την ομάδα των Πρασίνων θα συμφωνήσει ότι πρέπει να παρακολουθήσουμε από κοντά την κατάσταση αυτή στο Αφγανιστάν και να έχουμε μια πιο λεπτομερή συζήτηση για όλες τις απόψεις εκεί, για το πού βρισκόμαστε και για το τι είναι επιθυμητό, για το ποιες, είναι καλύτερες, ποιε θα πρέπει να είναι οι καλύτερες εξελίξεις για το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Νέιτς. Ζήτησε και πάλι το λόγο κυρία Λούνατσεκ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μετά τις παρεμβάσεις θα ήθελα να προσθέσω κάτι στην αρχική δική μου. Πρώτον, βεβαίως και καταλαβαίνω, καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα στο Αφγανιστάν. Δεν πρόκειται περί αυτού. Αυτό που τόνισα είναι ότι ε, θεώρησα ότι η διατύπωση που επελέγει μετά τις εκλογές έδωσε την εντύπωση ότι η κατάσταση θεωρεί το ε, πολύ πιο θετική από ό,τι στην πραγματικότητα. Όπως ξέρουμε τώρα, όπως έδειξαν τα πράγματα. Και θέλω να ξαναρωτήσω την Κομισιόν. Πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα. Πριν πάω εκεί όμως, ο κύριος Ομπιόλς Είπε επίσης πολύ σωστά ότι πάντοτε θα πρέπει να δούμε αν θα θεωρήσουμε μισοάδιο ή μισογεμάτο το ποτήρι. Το ξέρω αυτό. Αλλά ε, είναι και δική μας δουλειά. Αν υπάρξει αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να κρίνουμε τι θα μπορούσε να είχε πάει καλύτερα. Βεβαίω και συμφωνώ ότι ήταν δύσκολα τα πράγματα και η παρουσία μας εκεί και όλα. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να συμφωνήσω με την κυρία Νέιτς και κάποιους άλλους και εσείς το είπατε νομίζω κυρία Ομπιόλς ότι... Ε, καλό θα ήταν εμείς εδώ να περάσουμε σε ένα διαφορετικό στάδιο που θα συζητήσουμε τι είδους στρατηγικές αλλαγές θα απαιτηθούν στο Αφγανιστάν. Είναι σαφές τώρα ότι μόνο ο στρατός δεν βοηθάει. Και όλα αυτά τα χρόνια έγιναν πολύ λίγες επενδύσεις και οικονομικές και επιστώσεων, αλλά και σε ό,τι αφορά τους πόρους γενικότερα, στην κοινωνική σταθερότητα, την οικονομική σταθερότητα, ε, επενδύσεις ώστε ο λαός εκεί να καταλάβει ότι υπάρχει μια δυνατότητα νοικοδόμησης της χώρας. Πρέπει να γίνουν περισσότερα εκεί. Και αυτό πρέπει να το συζητήσουμε και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης, δεν θυμάμαι, με συγχωρείτε που ξέχασα το όνομά σας, ε, που είπατε ποια θα ήταν η εναλλακτική. Δεν λέω ότι δεν έπρεπε να έχουν γίνει εκλογές, όχι. Αλλά ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως Επιτροπή ΑΦΕΤ θα πρέπει να δούμε πώς έγινε η διαδικασία αυτή και τι μπορεί να γίνει. Και περνάω στην ερώτησή μου στην Κομισιόν. Αν υπάρξει άλλος γύρος, δεύτερος γύρος στις εκλογές αυτές, εσείς τι θα κάνετε, ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί για να ε, εξασφαλίσουμε ότι θα ε, γίνει σωστή εγγραφή των ε, ψηφιζόντων. Μπορεί, υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο να γίνει. Και τότε θα είναι πιο αξιόπιστες οι εκλογές. Δεν ξέρω. Ξέρω ότι είναι δύσκολες ερωτήσεις και ακόμα πιο δύσκολες οι απαντήσεις. Δεν ξέρω, ίσως έχετε απάντηση. Επίσης κάτι άλλο, δεν είναι μόνο η κοινωνική και, η κοινωνική και η οικονομική σταθερότητα και το θέμα των γυναικών όπως είπαν άλλοι, αλλά και το ζήτημα της δημιουργίας καλής διοίκησης. Και αυτό απαιτεί χρήματα και εκεί χρειάζεται να συζητήσουμε στρατηγικές που θα επικεντρώνονται περισσότερο στα πολιτικά ζητήματα σε αντιπαράθεση με τα στρατιωτικά, για να ενοικοδομηθεί το κράτος αυτό. Ωραία. Λίγη συζήτηση μεταξύ μας. Θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον δόκτωρα Μωράν και στην δόκτωρα Αρνό για τις ενδεχόμενες απαντήσεις, τις παρεμβάσεις και ερωτήσεις. Oh, uh, uh, um, Πρόεδρε, θα ήθελα να θίξω ορισμένα γενικότερα σημεία που ανέκυψαν από τη συζήτηση. Ως προς τη διαδικασία που εξελίσσεται, δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτά που συνέβησαν τις τελευταίες εβδομάδες. Υπάρχει η Εκλογική Επιτροπή Παραπώνων, Προσφυγών, ε, η οποία πλαισιώνεται και από διεθνείς εμπειρογνώμονες με πολύ μεγάλη αξιοπιστία και υποστήριξη από τη διεθνή κοινότητα. Επιτελεί την εργασία της λοιπόν, δηλαδή εξετάζει όλες τις εγγεγραμμένες πρόσφυγες και τις, εξετάζει εις βάθος έτσι ώστε να έχουμε καλύτερο ποιοτικά αποτέλεσμα μετά τον πρώτο γύρο της εκλογικής διαδικασίας. Θα χρειαστούμε μερικές εβδομάδες πριν λήξει αυτή η εργασία. Ε, ε, το δεύτερο είναι ότι η τελική έκθεση της Επιτροπής Παρατηρητών, όπως είπε και το αξιότιμο μέλος, θα συνταχθεί τον Οκτώβριο. Τώρα τι θα γίνει στο δεύτερο γύρο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να εικάσουμε κατά πόσο θα υπάρξει όχι δεύτερος γύρος και θα είναι πολύ δύσκολο να αποφανθούμε με βάση το input που έχουμε, ξέρουμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση και η Επίτροπος θα δει την κατάσταση in situ. Δεν ξέρω κατά πόσο ο Ρίτσαρτ Χόλμπρουκ αναφέρθηκε για έναν ενδεχόμενο δεύτερο γύρο. Υπάρχουν εικασίες, αλλά έχουμε πολλά ε, ενδεχόμενα αποτελέσματα. Η κυρία Λούνατσεκ ρώτησε κατά πόσο μπορούν οι πολίτες να συνεργαστούν. Υπάρχουν πολλές ε, δυνατότητες. Ο δόκτωρ Αμπτούλα ήταν υπουργός εξωτερικών υπό την κυβέρνηση Καρζάη, άρα ενδεχομένως να διανοίγονται και τέτοιες δυνατότητες, ε, ανεξάρτητα από την κυβέρνηση που θα ανακύψει. Επίσης, ε, ακούστηκαν πολλά σχόλια από τον δόκτωρα Αμπτούλα που έδειχναν ε, μετριοφρόση, που μάλλον ε, ήταν μετριοπαθή σχόλια. Αλλά δεν θα πρέπει να προβούμε σε εικασίες. Εάν γίνει δεύτερος γύρος, θα, ξέρουν, θα το ξέρουμε σε λίγες εβδομάδες. Αυτό, Αυτό που έχει σημασία είναι να έχουμε τα καλύτερα δυνατά ποιοτικά αποτελέσματα με βάση τις προϋπάρχουσες συνθήκες και η Εκλογική Επιτροπή Προσφυγών κάνει ό,τι μπορεί. Τώρα, προχωρώντας με τη νέα κυβέρνηση, οποιαδήποτε και να είναι και υπό την αιγίδα του οποιοδήποτε, θα αντιμετωπίσει μεγάλες ε, προκλήσεις και εμείς θα αντιμετωπίσουμε προκλήσεις διότι οι ΙΠΑ άλλαξαν τη στάση τους Ε, είναι υπέρ της αυγανοποίησης του κράτους. Ο ε, στρατηγός Μακρίσταλ και άλλοι διαβλέπουν μια διαφορετική δυνατότητα, δηλαδή η κατάσταση διαφέρει από τα τελευταία τρία-τέσσερα χρόνια. Βεβαίω, δεν ήμασταν πάντα επιτυχείς, αλλά τώρα έχουμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε με μια διαφανή κυβέρνηση έτσι ώστε να φτάσει αυτή η χώρα σε μια σταθερότητα και να υπόσχεται περισσότερα στους ανθρώπους μακροχρόνια, στους πολίτες μακροχρόνια έτσι ώστε να λάβουμε υπόψη και τη δέσμευση ασφάλειας που έχουμε αναλάβει έναντι αυτής της χώρας με τα μέχρι τώρα ε, τραγικά αποτελέσματα. Ε, ένας βουλευτής αναφέρθηκε σε αυτό το ζήτημα στις τραγικές απώλειες ως προς τις ε, έξωθεν συμβάσεις ε, δεν διαδραμάτισαν ρόλο. Επειδή εμείς είμαστε μεγάλοι δωρητές, θα ήθελα να πω ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Δηλαδή το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προωθήσουμε τον επιχειρηματικό κόσμο και τους κατασκευαστές εκεί. Τώρα το Πακιστάν είναι μια άλλη συζήτηση, ελπίζω να γίνει αυτή η συζήτηση. Μας ε, μιλήσατε για τη θέση του Πακιστάν. Αναμφίβολα, οι πακιστανικές στρατιωτικές δυνάμεις, οι ένοπλες δυνάμεις προσπαθούν να ελέγξουν τις ε, φυλές και ιδιαίτερα τους φονταμενταλιστές και τους Ταλιμπάν. Το τελευταίο σημείο που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι εμείς στην Επιτροπή θα θεωρούσαμε ευπρόσδεκτες μελλοντικές συζητήσεις για το Αφγανιστάν θα θέλουμε να αυξήσουμε την υποστήριξή μας για να σταθεροποιηθεί αυτή η χώρα τα επόμενα χρόνια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο υπ' αυτή του την ιδιότητα. Η Επίτροπος, αν ε, παρευρίσκεται ε, εδώ θα έλεγε ακριβώς το ίδιο. Βερονίκ, θες να προσθέσεις κάτι. Ευχαριστώ πολύ, αν μου επιτρέπετε σχετικά με την επιθυμία του κυρίου Όκελς να έχουμε τον κύριο Σέκουι και τον κύριο Μοριόν. Ο κύριο Σέκουι και ο κύριος Μπίλτ είναι στο Αφγανιστάν και ο κύριος Μοριόν επιστρέφει, είναι καθοδόν. Δεν ξέρουμε λοιπόν πόσο χρόνο θα διασκέσει η άλλη επίσκεψη. Δεν μπορώ να μιλήσω για τον κύριο Μοριό εφόσον οι αποστολέ μα ε, είναι ε, ξεχωριστές. Ίσως ε, η κυρία Νέη, ο κύριο Σαλαφράγκα ξέρουν κάτι. Είδαμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα αλλά ποτέ ένας επικεφαλής αποστολής δεν χρησιμοποίησε τις λέξεις free and fair, ελεύθερες και δίκαιες εκλογές. Τα πράγματα δεν είναι ποτέ λευμα, άσπρα ή μαύρα, είναι μια διαδικασία. Όπως το είπε η κυρία το ειπε η κυρια νειτσα μας ζητούν να πούμε ότι ε, αν ε, κάποιος έχει εκλεγεί. Εμείς δεν είμαστε εδώ για να επικυρώσουμε αποτελέσματα. Δεν, είναι αυτή η δουλειά μας. Όλοι συγκεντρώνονται στην ημέρα των εκλογών. Υπάρχει όμως όλη η διαδικασία πριν και όλη η διαδικασία μετά. Ε, βεβαίως είναι λιγότερο ορατά τα πράγματα εκεί και θα ήθελα να Αναφέροντας τον κύριο Μοριγιόν και να απαντήσω στην κυρία Λούνατσεκ, νομίζω ότι αυτό που θέλησε να πει, ερμηνεύω τα λόγια του, είναι ότι αυτό που ανακούφισε όλο τον κόσμο είναι ότι πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές. Πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές ενώ όλοι περίμεναν τα χειρότερα και όπως είπε ο κύριος Αταλμαντάλ και ο κύριος Αλαφράγκα, ε, κάπως ανακουφιστήκαμε επειδή οι ομάδες μας ε, κυρίως Ε, δεν υπέφεραν άμεσα, παρόλο που η κατάσταση ήταν πάρα πολύ δύσκολη και υπάρχουν πάρα πολλοί στρατιωτικοί που βρήκαν το θάνατο και η αστυνομία, η Αφγανική έκανε πολύ καλή δουλειά για, να, για την προστασία. Δεν είμαστε εδώ για να επικυρώσουμε αποτελέσματα, ίσως α, ε, περιμέναμε κάτι διαφορετικό από την αποστολή ίσως. Και κύριε Αυναντσέκ, όταν βλέπουμε τη διατύπωση λέμε ότι είναι λογικό το, το νομοθετικό πλαίσιο ότι έχουμε ε, κάτι το θετικό και το γεγονός ότι έλαβαν χώρα οι εκλογές είναι σημαντικό ε, για σχετικά μία από τις ε, κριτικές αρκετά οξίες που έκανε ο κύριος Μοριγιόν στην, στο ανακοινοθέν τύπου του είναι για την κατάσταση των γυναικών. Δύο πράγματα. Από τότε που η Επίτροπος Φεραίρο Βάλνερ έχει αυτό το χαρτοφυλάκιο και μας έδωσε οδηγίες και αυτό είναι που γίνεται τώρα, να έχουμε κάποιον στην αποστολή που να μελετά ιδιαίτερα το θέμα των γυναικών και στην ομοθεσία και στην ε, ψηφοφορία σε εκλογές στο Αφγανιστάν. Αυτό είναι, καταστροφή διότι δεν έχουμε αρκετέ και δεν έχουμε αρκετέ ψηφοφόρους. Ο κύριος Μέγερ ανέφερε επίσης ε, ε, το νόμο ΣΥΑ που είναι μια πολύ κακή έκπληξη. Ένα πρόβλημα. Αυτό το οποίο πρέπει να πω είναι ότι έχουμε ε, συνεργασία με την UNICEF στο Αφγανιστάν. Η κυρία Νέιτς εξήγησε ότι έχουμε επαφές με πάρα πολύ κόσμο. Η UNICEF έχει ειδικά προγράμματα. Προσπαθήσαμε λοιπόν να συνεργαστούμε με τη UNICEF. Αλλά ε, επίσης επαναλαμβάνω το ότι ήταν εξαίρεστες οι περιστάσεις. Θα ήθελα να κλείσω ε, με αυτό το οποίο είπανε πολλοί και ο κύριος Πλεύρης ότι πρέπει να περιμένουμε τα τελικά αποτελέσματα των εκλογών και, δεν θα, και θα πρέπει να μπορέσει η Επιτροπή Προσφυγών να κάνει τη δουλειά της. Δεν μπορούμε να κάνουμε προγνωστικά, αλλά είναι προφανές ότι για την ώρα έχουμε 2.030 ε, προσφυγές και 618 που θεωρούνται πολύ σοβαρές περιπτώσεις. Διαρωτώμεθα όλοι αν θα μπορέσουμε να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα της 21ης Σεπτεμβρίου, την προθεσμία αυτή. Ίσως να υπάρξει κάποια καθυστέρηση, αλλά για την ώρα αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να περιμένουμε και να προσποθήσουμε να καλμάρουμε τα πράγματα και να μην θεωρηθεί ότι αναμειγνιόμαστε στο πολιτικό παιχνίδι. Σας ευχαριστώ για τις ε, τελευταίες αυτές παρεμβάσεις από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα ήθελα να σας υποβάλω ορισμένες προτάσεις για τη συνέχεια αυτών των συζητήσεων. Νομίζω ότι υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον, αυτό κατέδειξαν οι διάφορες παρεμβάσεις και γι' αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει και στο μέλλον. Αύριο θα έρθω σε επαφή με τον πρέσβη Σέκουι που επιστρέφει από την Καμπούλ μετά από αυτή την επικοδομητική συζήτηση για να το ρωτήσω τι προτίθεται να κάνει μέχρι το τέλος του μήνα. Μέσα στα πλαίσια μιας συνάντησης στην οποία, την οποία δεν μπόρεσε να προωθήσει μέχρι τώρα λόγω ε, ανηλυμένων υποχρεώσεων. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα μας διαβάσει πολλές πληροφορίες και θα μπορέσουμε να εμβαθύνουμε το όλο ζήτημα. Ελπίζω να γίνει κατά τις, ε, μία από τις προσεχείς συνεδριάσεις προς το τέλος του μήνα. Στις 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου προβλέπεται μία συνεδρία στις Βρυξέλλες, επίσης στις 15 Σεπτεμβρίου στη, στο Στρασβούργο. Αν θέλετε μπορείτε να τις καταγράψετε αυτές οι ημερομηνίες. Ο Υπουργός Μπίλτ επίσης βρέθηκε στην ε, Καμπούλ, γι' αυτό και ο πρέσβης Σέκουι δεν είναι εδώ ε, μαζί μας. Ήθελε να τον υποδεχτεί in loco. Και στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων αυτό το Σαββατοκύριακο θα ασχοληθεί με το όλο θέμα και σε μία επόμενη φάση θα μας ε, μιλήσει για τα νέα δεδομένα όπως διαγράφονται. Επίσης θα ήθελα να καλέσω τον πρέσβη Σέκουι μέχρι το τέλος του μήνα να μας ενημερώσει επί του θέματος έτσι ώστε να μας ε, μιλήσει για τις ενδεχόμενες εξελίξεις στο Αφγανιστάν και Πακιστάν και να ζητήσουμε από τον στρατηγό Μοριγιόν να συναντηθεί μαζί μας σε μια κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Ανάπτυξης, διότι το Αφγανιστάν είναι μια ευαίσθητη περιοχή και έτσι θα έχουμε ένα σαφές πλαίσιο και θα ξέρουμε πώς προωθήθηκαν, πώς διενεργήθηκαν αυτές οι εκλογές, αν έληξε η εκλογική διαδικασία, αν θα χρειαστεί δεύτερος γύρος ή κατά πόσο αυτό το πολιτικό μάγμα δεν έχει επαρκώς οριστεί. Αυτές είναι οι ενδείξεις που έχουμε μέχρι τούδε. Ελπίζω να συμφωνείτε. Ως προς το πρόγραμμα που σας προανακοίνωσα, θα ήθελα να πω ότι μετά την, ε, τις εργασίες μας, ε, τις, ως ΑΦΕΤ, θα συναντηθούμε ως συντονιστές και ως διευρυμένο Προεδρείο. Άρα, ε, ε, λίγη συνεδρίαση της ΑΦΕΤ και θα ήθελα οι, αυτοί που δεν είναι άμεσα ενδιαφερόμενοι να αποχωρήσουν από την αίθουσα έτσι ώστε να αρχίσουμε με τις εργασίες του διευρυμένου Προεδρείου και του Διευρωμένου ε, Προεδρείου και των συντονιστών. Διακόπτουμε για λίγα λεπτά. Σας ευχαριστώ και θα ξαναειδωθούμε στις 15 Σεπτεμβρίου στο Στρασβούργο.